Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Με συγχωρείτε, αλλά Μόλις έκλεισε η ψηφοφορία. Έχετε κάποιο πρόβλημα με την κάρτα σας. Κυρία μου, έχετε κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημα. Ωραία, θα κοιτάξουμε να το επιδιορθώσουμε. 16. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. 13, με συγχωρείτε. 13, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1, παράγραφος 33, 31, άρχεται ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Συνεχίζεται να ψηφίζεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 12, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψήφισμα για τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων. Τροπολογία 1, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα, ονομαστική κλίση, στο σύνολό του, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο, επόμενη ψηφοφορία, αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού, ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική κλίση άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Επόμενο θέμα προς ψηφοφορία. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού μόλιβδο και ενώσει του. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για να επαληθεύσουμε. Πέρας. 3-5-3 ήταν η πλειοψηφία που χρειαζόμαστε και όπως βλέπετε ψηφίστηκε με 394 ψήφους υπέρ. Άρα ε, περνάει. Επόμενη εκθεσή στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τερματισμό τη πρακτική ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4, ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21ο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Πρώτο κατα αποχε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική Α. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική J, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. We can now move... Και τώρα πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή ΙΝΤΑ διαδικασίες αυτοποιημένης λήψης αποφάσεων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4, υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 5, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Αιτιολογική D. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ. Αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. επόμενο διαπραγματευτική εντολή για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράγραφος 2, σημείο 6, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ονομαστική κλίση μάλλον. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10, υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 14, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 14, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παραγραφός 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33, τοπολογία 1, υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε διότι εγώ δεν πρόσεξα αρκετά. Με συγχωρείτε. Παράγραφος 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξεκάθαρη έγκριση. 47 Τροπολογία 4, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία στο εδάφιο 50. Ο κύριος Γκούσμο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνουμε ότι η γενική συλλογιστική της έκθεσης είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, όπως γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, η υλοποίηση των όσων συμφωνηθούν με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ε, διαθετήσει και μια σειρά από προβλήματα στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών που εδώ και δεκαετίες διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με βασικές υπηρεσίες, συμβάσεις εργασία ή μισθώσεις ακινήτων. Εδώ λοιπόν ε, θέλουμε μια προφορική τροπολογία που να προστατεύει τον αυτόματη διευθέτηση και ομαλοποίηση, εξομάλυνση μάλλον της ε, κατάστασης αυτών των πολιτών και να εγκριθεί η ιδιότητα της κατοικίας τους. Αυτή είναι η τροπολογία μας. Ζητούμε την αυτόματη έγκριση μόνιμων θεωρήσεων διαμονής σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 30 Ιανουαρίου 2020 με εγγραφά ε, τυπωμένα τα οποία να αποδεικνύουν την κατοικία τους. Αυτά αφορούν το άρθρο 50, το σημείο 50 του ψηφίσματος. Πρόεδρος, το βασικό μέρος της ε, τροπολογίας αυτής είναι η τελευταία πρόταση, το προφορικό τμήμα της τροπολογίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την τροπολογία? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ κατά. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ συνάδελφοι, ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Να ελέγξουμε για την τροπολογία 2, παράγραφος 66, πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 77, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 78 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία Πέρα. εγκρίνεται 81 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία πέρας αυτής εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πράγματος 87 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 88 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 89 σε τρία τμήματα. Όλα ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτης έκθεση 2018 του κυρίου ε, Μαυρίδη. Δύο, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική κλίση. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Αρχικού κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν μπόρεσα να δω Οπότε θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ επί της παραγράφου 6 πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 υπέρ, κατά, αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ με τις κάρτες σας. Ψηφίζουμε με τις παραγράφου 12, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 με ονομαστική Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε επί του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 22, πρώτο τμήμα, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 με ονομαστική κλίση. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 2 στην παράγραφο 34. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23. Με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Συγγνώμη, πρέπει να το ξανακάνουμε είχαμε ένα προβληματάκι. Υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι. Θα σας ε, τα διαβάσω. Ψηφίζουμε επί 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και περνάμε στη ψηφοφορία Επί τη τροπολογία 25 με ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στην παράγραφο 44. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Θα το ε, επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί της τροπολογίας 4 στην παράγραφο 44. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αν μου ζητήσετε μπορούμε να το ελέγξουμε βεβαίως. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 15D. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 16D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 με ονομαστική κλίση. άσχετη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Okay, I need to redo that because it's showing um, Amendment 116D where we are voting on Amendment 26. Okay. Σας έδειχνε την ε, τροπολογία 16D ενώ ψηφίζαμε για την 26. Μπορούμε να το ξαναρχίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε επιστροπολογίες 26 με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. That is rejected. We... Απορρίπτεται. Ετουλογική σκέψη C1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 στην ετουλογική σκέψη M υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην ψηφοφορία επί του ψηφίσματος στο σύνολό του με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Παράνομο ζω... Ε, εμπόριο ζώων συντροφιάς. Παράγραφος 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, στην παράγραφο 10, με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1, στην παράγραφο 36, υπέρ, κατά, Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι δεν συγκεντρώνεστε. Περνάμε ξανά. Παράγραφος 36, τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Συντολική σκέψη D. Υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε κιόλα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί τη τροπολογία 5 στην εντολική σκέψη D. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκτρολογική σκέψη M, τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε κι αυτό. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 6, πέραση τη ψηφοφορία. εγκρίνεται και με μεγάλη διαφορά. Περνάμε στη ψηφοφορία επί του ψηφίσματο στο σύνολο με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται, συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ πολύ και περνάμε σε επεξηγήσει ψήφου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω. Περνάμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Amint Σας παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα όσοι το επιθυμείτε για να μπορούμε να περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτη επεξηγήση ψήφου αφορά την ψηφοφορία για τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Η Ραφαέλα Ζαμέρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Dear colleagues, there are 80. Συναδελφοί, 80 είναι οι ομιλητές για την επόμενη ώρα, μια μισή ώρα, οπότε παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ραφαέλα, έχετε το λόγο. Συνάδελφοι, σήμερα το πρωί ψήφισαμε υπέρ της συμφωνίας με το Βιετνάμ. Δεν ήταν κάτι το εύκολο, αλλά μετά από σκέψη αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ. Όμως η κατάσταση στη χώρα απέχει πολύ από το να είναι ιδανική. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτές οι συμφωνίες με το Βιετνάμ όχι μόνο θα βελτιώσουν τις εμπορικές σχέσεις με τη χώρα, επίσης θα αποτελέσουν μια πλατφόρμα διαλόγου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ωφεληθεί ο λαός της χώρας. Οι εταίροι μας θα έχουν στο το δυνατό επίπεδο περιβάλλον και δικαιώματα. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει εάν όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε να υπάρχει ευρύτερη υποστήριξη από όλες τις πολιτικές πτέρυγες για τέτοιες συμφωνίες. Κύριε Αουμπρή, από πλευράς Γκουε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μπράβο αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίσατε αυτή την Συμφωνία Ελευθέρων Συνεργού με το Βιετνάμ που δεν σέβεται τα δικαιώματα και το περιβάλλον για να ικανοποιήσετε τα λόμπι που σας κερνάνε σαμπάνια. Καταστροφή οικολογική. Για θα διευκολύνετε τα εμπορεύματα, αλλά θα καταστραφούν τα δάση, ε, θα καταστραφούν οι χαλιβουργίες, αλλά παρόλα αυτά εσείς ψηφίσατε πριν αυτή της συμφωνίας που κάνει κακό στο κλίμα. Κοινωνικό σκάνδαλο. Εκμετάλλευση. Εξυπηρετείτε τον αυταρχισμό και την παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού. Φυλακίζονται στη χώρα συνδικαλιστές και αντιφρονούντες, άρα θα πρέπει να σκεφτείτε τις καταστροφικές συνέπειες. Αλλιώς είστε υπεύθυνοι και ακόμα χειρότερο είσαστε κοινικοί. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Φιτζέρλ ε, ε, για το PP. οπότε τώρα θα έχουμε απασχόληση εμπορικές συναλλαγές με την ε, χώρα. Χρειάζεται απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε την καινοτομία και την απασχόληση. Αν κλείσουμε την πόρτα, δεν βελτιώνουμε την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για την κλιματική αλλαγή. Ο ΙΕ και η ΜΚΟ αναγνώρισαν ότι είναι θετικό βήμα και υπάρχει κεφάλαιο για δικαιώματα στην συμφωνία και μεταφέρονται και οι διατάξεις του ILO. Βεβαίω θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται και να παρακολουθήσουμε συνεχώς την εφαρμογή της συμφωνίας. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τους δώσουμε προοπτική για νέους χώρους και έτσι να μεταφέρουμε τις ε, αξίες και τις ιδέες μας ως Ευρώπη. Κυρία Σόιντροβε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ψήφισα υπέρ αυτής της ε, συμφωνίας. μάλλον ψήφισα υπέρ της συμφωνίας, διότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις σχέσεις μας με αυτή την περιοχή του κόσμου. Ε, είναι καλό να προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα την, τον κόσμο απασχόλησης και την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς η συμφωνία δεν είναι αρκετά ισχυρή βέβαια για να επιτρέψει στην ε, κυβέρνηση να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Και το Βιετνάμ καθώς και η Βιετναμαζική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατευτούν πραγματικά οι ελευθερίες των πολιτών και τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρου Βόντρε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Προ, α, τα Εγώ υπερψήφισα και δεν μπορώ να καταλάβω την ιστερία που ε, βλέπω στο άλλο άκρο εδώ του ημικυκλίου. Μου δείχνει ότι μάλλον σωστά ψήφισα. Γιατί εγώ θυμάμαι την περίοδο του κομμουνισμού. Κάποιες φορές γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταχειρίζεται κανείς ε, ε, ή να διαμορφώνει μια στάση απέναντι σε καθεστώτα που φυλακίζουν αντιφρονούντες. Και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση, το Βιετνάμ. Θεωρώ όμως ότι το εμπόριο μπορεί να ε, βοηθήσει τα πράγματα, να βελτιωθούν τα πράγματα. Γι' αυτό και θέλω να καλέσω την Κομισιόν πάντοτε στις συνομιλίες της με το Βιετνάμ και στις μελέτες επιπτώσεων να λαμβάνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μπομπάχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το κοινοβούλιο σα ενέκρινε για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φοντερ Λάιεν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Αυτή η συμφωνία είναι επιζήμια για τη δημοκρατία, του εργαζομένου και το περιβάλλον. Επιζήμια για τη δημοκρατία, γιατί αυτή η δημοκρατία με το αυταρχικό και κατασταλτικό καθεστώ του Βιετνάμ ε, θα επιτρέψει να θριαμβεύσουν τα δικαστήρια επίλυση διαφορών που συνήθω ε, δίνουν προτεραιότητα στι πολυεθνικέ ε, σε σχέση με του λαού. Είναι επιζήμιο για του εργαζομένου, διότι μιλάμε για 2 εκατομμύρια εργαζόμενων στην κλωστοεφαντουργία που ζουν σε συνθήκε κοινωνικού dumping. Αυτή η συμφωνία θα συνεχίσει την εκμετάλλευσή του από τι πολυεθνικές, από τις πολυεθνικές και την κυβερνήσει του. Τι γίνεται με τι συμβάσει του ε, Οργανισμού Εργασία και ε, των όσων θα έπρεπε να ισχύουν ε, διεθνώ. Επίση για το περιβάλλον είναι επιζήμια, διότι δεν επιτρέπει να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι των διεθνών συμφωνιών για το περιβάλλον. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα θα αυξηθούν ε, εξαιτία αυτών των ελεύθερων συναλλαγών. Γι' αυτό καταψηφίζω και μάλιστα ε, έντονα την ε, κακή αυτή συμφωνία. Ευχαριστούμε και τώρα Μίλαν Πέρες για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών κυρίω, είναι αξίε οι οποίε βρίσκονται στα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνή συνεργασία τελικά υποκαθίσταται από τον λαϊκισμό ε, και τον εθνικισμό τη τάση εθνικού προστατευτισμού παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται λοιπόν τι συμφωνίε αυτέ με τι τρίτε χώρε. Δυστυχώ εδώ υπάρχει μια ε, μειοψηφία που πιστεύει ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τα χαμηλά πρότυπα, τα χαμηλά δημοκρατικά πρότυπα στο Βιετνάμ. Εγώ γι' αυτό ε, καταψήφισα την συμφωνία αυτή, διότι δεν θα επιτρέψουμε να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με τέτοιε συμφωνίε. Πρέπει να είμαστε πιο ευθύ, πιο απαιτητικοί και αυστηρότεροι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση στα χέρια τη Κίνα και των ΗΠΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ έχει βελτιωθεί τόσο πολύ, ε, τότε γιατί η δημοσιογράφος Φαμ Σιντούν έχει συλληφθεί και βρίσκεται στη φυλακή με ποινές, με κατηγορίες από την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο κατηγορείται. Ε, εδώ ε, το Κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας, ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι αν δεν συνάψουμε σχέσεις μαζί τους πώς θα βελτιωθούν τα δικαιώματά τους. Αυτό πραγματικά είναι πρόκληση για το χιλιάδε ανθρώπου, εκατοντάδε ανθρώπου που μα ζήτησαν να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία όταν επικοινωνήσαν μαζί μα. Του προδίδουμε τώρα. Εγώ λοιπόν γι' αυτό καταψήφισα την ε, συμφωνία αυτή. Και για το συγκεκριμένο λόγο ε, και γιατί δείξαμε ότι είμαστε ε, μια ομάδα από υποκριτέ στην ουσία. Πέρασε στι 15 Ιανουαρίου ένα ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και Είπαμε ότι θα έχουμε εμπορικέ συμφωνίε με αυστηρέ ε, ρήτρε για την βιώσιμη ανάπτυξη και την Συμφωνία των Παρισίων. Εδώ κάναμε το αντιδιωματικά αντίθετο. Ντροπή μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπελαμία, εκ μέρου του ΕΛΚ. Συνάδελφοι, η ψήφιση της συμφωνίας ήταν ε, ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο. με όλες τις ενστάσεις που αναφέρθηκαν που ήταν ε, βάσιμες και κυρίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ενισχυτικά στο Βιετνάμ. Αλλά ε, αυτά δεν έπεσαν στο κενό. Θέλουμε σαν αλλαγές με το Βιετνάμ που είναι ήδη εταίρος της Ένωσης. Είναι υπέρ του Βιετνάμ. Είναι χώρα που έχει εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με μας. Άρα θα πρέπει αυτό να κάνουμε. Θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρο να έρθουν κοντά μας και να αγκαλιάσουν αυτούς τους στόχους, τους οικολογικούς, τους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό το κάνουμε με τις εμπορικές αλλαγέ σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς ε, που διέπονται από την αμοιβαιότητα. Με αυτή τη συμφωνία ε, κάνουμε βήματα θετικά και αν δεν ε, συναυθεί αυτή η συμφωνία, τότε θα προσεγγίσει το Βιετνάμ την Κίνα. Ε, δεν το θέλουμε αυτό. Ε, σε αυτό είναι παρέτηση που δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μπελαμή. Και τώρα ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <coughs> Ψηφίσα κατά τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών γιατί νομίζω ότι θα είναι αρνητικέ οι συνέπειες για την οικονομία και την απασχόληση ήδη έχουμε πάρα πολλά τέτοια προϊόντα χαμηλού κόστου στην Ένωση, γι' αυτό και είναι πλεοναστική 27 ε, δις το 18. Ε, αυτή η κατάργηση και μείωση των δασμών θα κάνει το δικό μας έλλειμμα ακόμα μεγαλύτερο. Θα έχουμε επίσης με την κατάσταση επιχειρήσεων. Επίσης πρόκειται για μια κομμουνιστική δημοκρατία. Δεν σέβεται τα δικαιώματα ούτε περιβάλλον. Επομένως ε, ε, είναι υποκριτικό να θεωρήσουμε ότι έτσι τα πράγματα όλα θα γίνουν ρόδινα. Και για άλλη μία φορά προδίδει η Ένωση της αξίας που υποτίθεται ότι σέβεται. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με το Βιετνάμ είναι η πρώτη τέτοια ε, συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αναπτυσσόμενη χώρα. Το Βιετνάμ βεβαίω δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ιδανικό εταίρο. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να εξασφαλίσει κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Όμω για αναπτυσσόμενη χώρα το Βιετνάμ έχει αναλάβει πολύ σημαντικέ δεσμεύσει. Και θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή θα φέρει ευκαιρίε τόσο για, Ευρω... για του Ευρωπαίου και του Βιετναμέζου εργαζόμενου και τι επιχειρήσει. Και είναι σημαντικό το ότι προβλέπονται υψηλής ποιότητας κανόνες, όπως είναι για παράδειγμα η κύρωση των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Άρα η συμφωνία αυτή έχει και πολιτική σημασία γιατί αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Βιετνάμ να μην βασίζεται μόνο στις εμπορικές του σχέσεις με την ε, Κίνα. Θα συνεχίσουμε και θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν, είναι, δεν πρόκειται για το τέλος της διαδρομής. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και το διάλογό μας κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίηση τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλούν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστήριξα το ψήφισμα και τη συμφωνία με το Βιετνάμ, γιατί πιστεύω ότι οι εμπορικέ συμφωνίε αποτελούν ευκαιρία για να μπορέσει κανεί να δραστηριοποιηθεί σε όλου του τομεί, περιβάλλον, κοινωνικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εμπορικέ συμφωνίε ωφελούν του καταναλωτέ, τι επιχειρήσει και δημιουργούν θέσει εργασία και στι δύο πλευρέ. Αναγνωρίζω ότι το Βιετνάμ δεν είναι ιδανική χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμω μέσω τη συμμετοχή και των επαφών που θα έχουμε χάρη σε αυτή τη συμφωνία μέσω των επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται εκεί, νομίζω ότι θα υπάρχουν ωφέλη και πλεονεκτήματα και για επιχειρήσει και του καταναλωτέ και στι δύο πλευρέ. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ε, εφαρμογή και υλοποίηση αυτή τη συμφωνία, ιδίω όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω μια συμφωνία εμπορική ε, που θα βασίζεται σε κανόνες, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το να μην υπήρχε μια τέτοια συμφωνία και πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές με το Βιετνάμ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βρετσιονόβα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Υποστήριξα το ψήφισμα και την έκθεση για τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Σε μια περίοδο θέσπισης νέων δασμών και εμπορικών πολέμων θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό το μήνυμα. Εγώ ως άνθρωπος που μεγάλωσα στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία βεβαίως ε, στάθμισα ε, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως θεωρώ ότι μέσω αυτής της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στα χέρια της ένα εργαλείο το οποίο θα της ε, επιτρέψει να βελτιωθεί η κατάσταση και ως προς το περιβάλλον. Και πέρα από την βελτίωση των εμπορικών σχέσεων, θεωρώ ότι και σε αυτού του τομεί θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε ε, βελτιώσεις. Από το ECR ο κύριος Ζαχραντήλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν εισηγητή για τις δύο αυτές συμφωνίες από το 2012 έως το 2019. Εγκατέλειψα τη θέση αυτή γιατί διαδόθηκαν εναντίον μου διάφορα ψεύδη από τους πράσινους και, τους, ε, και το κόμμα των πειρατών. Ότι δήθεν ήθελα να υπονομεύσω την ε, ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών με το Βιετνάμ. Δεν ίσχυε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον ενέκρινε τις συμφωνίες αυτές, διότι στέλνει το σωστό μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δείχνει ότι σε μια εποχή εμπορικών δασμών και προστατευτισμού υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ευχαριστώ ο Σον Κέλλη εκ μέρους του ΕΛΚ. Uh, Ευχαριστώ. Υποστήριξα τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Ω μόνιμο εισηγητή του ΕΛΚ για την περιοχή τη Νοτιοανατολική Ασία και επειδή έχω υποστηρίξει και τη Συμφωνία ε, με τη Σιγκαπούρη, γνωρίζω πόσο μεγάλε δυνατότητε έχουν αυτέ οι συμφωνίε να ενισχύσουν τι εμπορικέ μα σχέσει με αυτέ τι περιοχέ, τι χώρε αυτέ τη περιοχή. Για το περιβάλλον και ένα καλύτερο, ασφαλέστερο ε, χώρο για τι επενδύσει. Η Συμφωνία ανοίγει νέε προοπτικέ, κυρίω με την εξάπληψη 99% ε, των φραγμών και δεσμολογικών φραγμών, μη δεσμολογικών μάλλον φραγμών. Ε, για τα ε, προϊόντα, για τα τρόφιμα, το γάλα, το κρέας πουλερικών και το χείριο υπάρχουν μεγάλες διευκολύνσεις χάρη σε αυτή τη συμφωνία και, προς, και για τις εξαγωγές μας προς το Βιετνάμ. Ελπίζω λοιπόν να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστούμε. Και τώρα... Ο λόγος και πάλι στο συνάδελφο που δεν ακούστηκε καλά η παρέμβασή της λόγω του θορύβου στην αίθουσα. Okay. Συγγνώμη, συναδέλφοι, το πρωί ε, ψηφίσαμε υπέρ τη διαδικ... της συμφωνία με το Βιετνάμ. Δεν ήταν απλή διαδικασία, αλλά μετά από προσεκτική ε, μελέτη τη κατάσταση αποφάσισα να υπερψηφίσω. Δεν είναι ιδανική η συμφωνία. Η Βιετναμέζικη όμω κυβέρνηση έχει κάνει δεσμεύσει προ τη σωστή κατεύθυνση. Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και αυτή τη προστασία των επενδύσεων θα βελτιώσουν όχι μόνο τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ, αλλά θα δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για να συνεχιστεί ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Βιετναμέζικη ε, ε, πλευρά και να μοφεληθούν οι πολίτε του Βιετνάμ. Η εμπορική μα εταιρική σχέση θα επιτρέψει τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα να παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. Θέλω λοιπόν να συστήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο στόχων και διαφανών κριτηρίων για να χρησιμοποιηθούν ω ε, πύχη για να προχωρήσουν προ αυτήν την κατεύθυνση οι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει όλε οι πολιτικέ πτέρυγε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν αυτή την κίνηση. Ευχαριστούμε. Και τώρα ολοκληρώνω το κατάλογο των αγορητών. Τρει Τρία αιτήματα παραμένουν για το επόμενο σημείο ε, εξήγηση για, ε, για το ψήφισμα της έκθεσης Μπουρζουά για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συνολογών, κυρία Ρούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ψήφο σε αυτή ήταν το και χθε εξηγήθηκε γιατί αντιβαίνει τελείω αυτή η συμφωνία με το ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή και για κάτι υπέρ της νέας συμφωνίας. Ε, δεν ήταν δυνατόν οι πράσινοι να ψηφίσουν αυτή την συμφωνία λόγω της κατάστασης δικαιωμάτων σε αυτή την αυταρχική χώρα. Αλλά επίσης δεν τηρεί η χώρα και όσα επιτάσσει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Υπάρχει πολύ αρνητική επίπτωση όσον αφορά την λαθραλία ε, και την παρανομιαλία γιατί έχει φάει πολλές κίτρινες κάρτες στο Βιετνάμ γιατί δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα όσον αφορά ε, την λαθραλία εδώ και λίγους μήνες προσπαθεί να συμμορφωθεί αλλά ακόμη παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες για το θέμα της αλίας. Με την έγκριση αυτής της συμφωνίας αυτό το σύστημα των κίτρινων καρτών το αποδυναμώνουμε. Επίσης αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε εισαγωγές ε, υποπροϊόντων αυτής της ε, λαθραλίας. Στάνισλαβ Πόλτσοκ για το Λαϊκό Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε γιατί προερχόμαστε από πρώην κομμουνιστικές χώρες. Τελικά ψήφισα υπέρ της συμφωνίας. Είναι πιο πολλά τα πλεονεκτήματα από τα μειονεκτήματα. πιο εύκολο είναι να τηρούνται κάποιοι κανόνες και να εμπορεύεται κανείς, γιατί αν δεν υπάρχουν κανόνες δεν μπορεί κανείς να επηρεάσει τα όσα γίνονται στη χώρα. Ήδη συνεργαζόμαστε με την χώρα και θεωρούμε ότι το εμπόριο δίνει δυνατότητες ούτω ώστε να υπάρξει συμμόρφωση για τα περιβαλλοντικά αλλά και τα εργασιακά. Και για αυτό ψηφίσαμε υπέρ. γόλας. Πολλά κοινά στοιχεία βλέπουμε για προηγούμενες συμφωνίες της ΣΥΤΑ με Ιαπωνία, Κορέα, Μερκοσούρ. Αυτές οι συμφωνίες έχουν τις ίδιες επιπτώσεις και συνεχώς κάνουμε το ίδιο λάθος δίθεν υπέρ του ελευθέρου εμπορίου ενώ ο κόσμος υποφέρει. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να μην λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Θα, δυστυχώς θα γίνουμε μάρτυρες της καταστροφής του κλίματος. Η δημόσια υγεία δεν προστατεύεται έτσι. Όλα για την παγκοσμιοποίηση γίνονται. και κάποιοι πλουτίζουν με τις εξαγωγές που γίνονται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων. Η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστήριξα την Συμφωνία προστασία των Επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ. Γιατί έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα από την προηγούμενη συμφωνία. Την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Διότι εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πέμπτο μεγαλύτερο επενδυτή στο Βιετνάμ. Είναι μεγάλο εταίρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά συνέπεια να προστατεύονται οι επενδυτέ και οι επενδύσεις τους στο Βιετνάμ και η συμφωνία αυτή θεσπίζει σαφείς κανόνες. Οι επενδύσεις ε, στο Βιετνάμ δημιουργούν νέε θέσει εργασία. Και θέλουμε το Βιετνάμ να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ε, οικονομικά, αλλά και ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία των πολιτών τους. Στην ε, Τσεχία ζουν περίπου 60.000 ε, Βιετναμέζοι. Η κατάστασή τους δεν είναι καθόλου εύκολη. Η συμφωνία όμως αυτή θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στη Βιετναμέζικη κυβέρνηση ώστε να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω το Βιετνάμ με συμπάθεια, διότι ήμουν ε, υπεύθυνο από τη Γαλλία ε, επί πέντε χρόνια για τι σχέσει με την Ανατολική Ασία. Εδώ λοιπόν εκτιμώ τι προσπάθειε τη χώρα αυτή να ξανασταθεί ξανά στα πόδια τη. Εδώ πρέπει να εργαστούμε όμω με αντικειμενικά δεδομένα και να πετύχουμε να ε, συσφίξουμε τι σχέσει μα με πολλέ χώρε του κόσμου. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τι διεθνεί σχέσει, κυρίω για τα ανθρώπινα δικαιώματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κραδένει σε κάθε περίπτωση. Εγώ καταψήφισα όμω τη συγκεκριμένη συμφωνία γιατί δεν ωφελεί του Ευρωπαίου, διότι διέπεται από τον αφιερωισμό των ελεύθερων συναλλαγών και ε, όχι για τα δικαιώματα των λαών. Δεν ε, θέλω να ε, Προσπογράψω σε καμία συμφωνία που ε, επιτρέπει την ε, επαναγκατάσταση βιομηχανιών εκτό Ευρώπη. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε η δικαιοσύνη, ε, η διατησία και η επίλυση διαφορών να περάσει στα χέρια των ιδιωτών σε σχέση με τη δημόσια δικαιοσύνη, την κρατική δικαιοσύνη. Γι' αυτό καταψήφισα το κείμενο αυτό για τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Με της, με το έργα κοινού ενδιαφέροντος, κυρία Ένστ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό και ε, κατά συνέπεια κατά του καταλόγου για τα έργα κοινού συμφέροντος. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτόν τον κατάλογο προβλέπεται ότι θα χρηματοδοθούν 50 ε, έργα ε, φυσικού αερίου και Πρόκειται για χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία ε, είναι ε, βλαπτικά για το περιβάλλον. Αν θέλουμε μέσω των, ε, συμφωνιών μας να προωθήσουμε το περιβάλλον, ε, θεωρώ ότι αυτή η, αυτό το ψήφισμα είναι πραγματικά ντροπή, διότι στην ουσία καταργούμε την ίδια τη Συμφωνία των Παρισίων διότι τελικά χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό έργα για ε, φυσικού αερίου. Δεν συμφωνούμε. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για μεθοριακά έργα. Για παράδειγμα, ηλιακή ενέργεια από την Ισπανία που θα μπορούσε να μεταφέρεται προς το βορρά της Ευρώπης ή έξυπνα δίκτυα τα οποία πράγματι θα, θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Αυτά, αυτά θα πρέπει να είναι οι στόχοι και αυτά δεν συμβαδίζουν με τα όσα προτείνονται εδώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα πάλι από την ΚΟΕ, κυρία Ομπρή, για ένα λεπτό. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις παρουσίασε με ε, πανηγυρισμούς την Πράσινη Συμφωνία, τώρα έχουμε ένα κατάλογο επενδύσεων που ηρωνικώς ε, αποκαλείται κοινού ενδιαφέροντος που υποτίθεται ότι αφορούν 32 έργα ε, που βασίζονται στο φυσικό αέριο. Για ποιο κοινό ενδιαφέρον μιλάτε, ε, κοινό όφελο, όταν θέλετε να στηρίξετε τη βιομηχανία φυσικού αερίου και το ε, φυσικό αέριο είναι 20% των διεθνών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Για ποιο κοινό ενδιαφέρον μιλάτε, όταν θέλετε να δώσετε 9 δι δημόσιων κομπηλίων για να προωθήσετε αυτά τα κλιματοκτόνα έργα. Και πώ το φυσικό αέριο που προέρχεται από την υδρορογμάτωση και καταστρέφει του υδροφόρου ορίζοντε, θα βοηθήσει τον πλανήτη και τι τοπικέ κοινότητε.